på Εξ Επιτροπής Γυναικών και Ελευθεριών θα ήθελα να σα καλωσορίσω στη σημερινή κοινή συνεδρίαση ανάμεσα στην Επιτροπή Γυναικών και Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Έχουμε δύο σημαντικότατα ζητήματα για τα οποία θα ψηφίσουμε σήμερα, αλλά θα πάρουμε με την αρχή σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης για την κοινή μας συνεδρίαση. Υπάρχουν ενστάσεις. Δεν έχω λάβει τίποτα, οπότε θεωρώ εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2, ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις σήμερα. Σημείο 3, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 13ης Ιουλίου, 2 Σεπτεμβρίου και 29ης Σεπτεμβρίου. Εάν δεν υποβάλλεται ενστάσεις πριν τη λήξη της σημερινή ε, συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο 4 λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Στις 25 Νοεμβρίου και όχι νωρίτερα, κάναμε άλλη μια κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών όπου οι δύο συναρμόδιοι εισηγητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και είχαν την ευκαιρία και είχατε και εσείς την ευκαιρία να τοποθετηθείτε για τις μελλοντικές εργασίες. Τώρα θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές. Η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ Μπάριο θα πάρει πρώτη το λόγο, παρακαλώ. Eh, Μάλιστα, πρωτού ψηφίσουμε. Θα ήθελα κάποια λόγια να αναφέρω. Το κείμενο είναι ένα καλό κείμενο, πιστεύω. Αποδεκτό, παρότι όλοι θα θέλαμε να είναι πιο φιλόδοξο και να πήγαινε πιο πέρα. Αλλά μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι είναι το μέγιστο που καταφέραμε να πετύχουμε. Και ευελπιστώ, πιστεύω ότι δεν εγκαταλείψαμε τον κυριότερο στόχο μας που ήταν η προστασία των θυμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω ότι εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο εκπρόσωποι των πολιτών και των θυμάτων που φοβούνται και υποφέρουν και έχουν δικαίωμα να ζουν σε ελευθερία και με ελπίδες Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα εμείς και πρέπει να υπερψηφίσουμε στην δική μας Κοινοβουλευτική Επίτροπη και να προχωρήσει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου αυτή η έκθεση. Γιατί αυτή είναι η φωνή του Κοινοβουλίου, έτσι αρθρώνεται. Πρέπει να την ακούσει το Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να προστατέψουμε τα θύματα και γι' αυτό εργαστήκαμε. Και δεν θα απεμπολίσουμε, δεν θα εγκαταλείψουμε αυτόν τον στόχο, που είναι ένας στόχος δίκαιος και θέλουμε εμείς και πιστεύουμε σε αυτόν τον στόχο και πιστεύουν σε αυτόν όλοι οι πολίτες. Ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στην εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Η κυρία Ρουμίρο έχει τον λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό είναι το τέλος ε, μιας ε, κοινοβουλευτικής πορείας ε, για αυτή την εντολή προστασίας που τόσα πολλά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εξέτασής της. Μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο τέρμα της διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο με ένα μείγμα γλυκό πικρό σε αυτό, ως αποτέλεσμα διότι οι πρωτοβουλίες όπως όλες οι πρωτοβουλίες πολλά πράγματα εγκαταλείπονται καθοδόν αλλά αντέξαμε και κρατήσαμε ως το τέλος την ανάγκη την κατεπίγουσα ανάγκη αυτού του μέσου διότι απομακρύνει εκείνους που επιτίθενται από τα θύματα και εκείνοι που ζητούν προστασία σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προστατευθούν. Σήμερα πιστεύουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα επικυρώσει αυτή την απόφαση, να δρομολογηθεί αυτό το μέσο με τέτοιο τρόπο ώστε κατεπηγόντως να λειτουργήσει. Διότι ήδη έχουμε διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο εμείς για αυτό το θέμα είναι ένα από τα μέσα που εγώ πιστεύω ότι θα δώσουν, θα τιμήσουν αυτό το κοινοβούλιο ως αποτέλεσμα έχοντας αναζητήσει εμείς τη συμφωνία κυρίως όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων και επιπλέον επειδή βγαίνει ε, εκφράζεται η ανάγκη για ένα θέμα που είναι κατεπήγον σήμερα στην Ευρώπη. Να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να προστατεύονται τα θύματα, όπου και αν βρίσκονται αυτά τα θύματα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η ευθύνη είναι στα χέρια του Συμβουλίου πια. Και ενθαρρύνουμε, προτρέπουμε το Συμβούλιο να εξετάσει μια και το Κοινοβούλιο όπως το εξέτασε με κατεπήγουσα διαδικασία να το κάνει και το Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει ώστε να μπορέσει να δρομολογηθεί αμέσως αυτό το μέσο ώστε τα θύματα να προστατεύονται το δυνατόν πιο νωρίς, πιο γοργά και να το εξετάσει με την διαδικασία του κατεπήγοντος στο Συμβούλιο και να φτάσουμε στην Ολομέλεια με τα καλά μαντάτα ότι το Συμβούλιο δίνει πράσινο φως και εγκρίνει. Ευχαριστώ όλους που κατέστησαν εφικτό και συνεργά για να φτάσουμε στο τέλος αυτής της πορείας με μια συμφωνία των ομάδων και με τη συνεργασία που ήταν πάρα πολύ αξιόλογη, ανεκτήμητη συνεργασία και για τις τροπολογίες όλων των ομάδων και όλων όσων εργάστηκαν από κοινού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρομέρο. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, ο κύριος Ντεμπορμπιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Βελγική Προεδρία ναι καθένα προσέδιδε και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οδηγία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Ήδη από τις 29 Σεπτεμβρίου από την ψηφοφορία προς Ανατολισμού εργαστήκαμε εντατικά ε, σε συνεργασία με τους εισηγητές για να καταλήξουμε σε συμφωνία και θα θέλαμε εξ ονόματος της Βελγικής Προεδρίας να ευχαριστήσουμε τους συνεισηγητές ε, για την συνεργασία τους. Ε, και τον σημειώνουμε την ισχυρή δέσμευση του Κοινοβουλίου ε, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας όπως προέκυψε από τις ε, διαπραγματεύσεις. Νομίζουμε ότι προσεγγίζουμε μια λύση αποδεκτή για τα δύο θεσμικά όργανα. Αυτό φάνηκε ήδη από το τελευταίο τριμερή διάλογο. Στο Συμβούλιο κάποιες αντιπροσωπείες είχαν κάποιες δυσκολίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του νομοθετήματος. Το προτινόμενο πεδίο εφαρμογής συζητήθηκε στις διαπραγματεύσεις και έτυχε παρκούς υποστήριξης ε, και από πλευράς του Κοινοβουλίου. Ε, σημειώθηκαν κάποιες εξελίξεις στα τελευταία στάδια ως προς την κοινή θέση του Συμβουλίου, δηλαδή η ομάδα των κρατών που δυσκολευόντουσαν με το πεδίο εφαρμογής ε, ε, ε, είδε τη θέση της να ενισχύεται και τελικά επιζητήθηκαν και βρέθηκαν λύσεις με τους συνεισηγητές για τις διάφορες πτυχές της πρότασης οδηγίας, όχι μόνο για το πεδίο εφαρμογής. Το Συμβούλιο τώρα για κάποιο χρονικό διάστημα θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και προφανώς θα λάβουμε δεόντως υπόψη την ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου θα λάβουμε υπόψη το μήνυμα που θέλει να αποστείλει προς το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε για το ενοποιημένο κείμενο. Τροπολογία 231 υπέρ παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη, μπορείτε να με προσθέσετε, γιατί δεν έχω την ηλεκτρονική μου κάρτα μαζί. Ναι, ναι, και ε, θα ψηφίσετε υπέρ αν το κάνω αυτό, έτσι, λέει αστειευόμενη πρόεδρος. Ε, πέρασε της ψηφοφορίας. 46. 47 υπέρ, 0 ε, ψήφι κατά και 5 αποχές. Συγχαρητήρια. σανόματος και των δύο επιτροπών θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεισηγητές μας και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, όλα τα μέλη και των δύο επιτροπών για την λιαναγκαστή συνεργασία που είχαμε. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο. Επίσης ένα κοινό σημείο για τις δύο επιτροπές. Πρόκειται για την πρόταση οδηγίας για την εμπορία ανθρώπων. Και εδώ έχουμε δύο συνεισηγητές, ε, συνεισηγήτριες μάλλον, μία από την Επιτροπή Γυναικών και μία από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η κυρία Μπάουερ είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Γυναικών, αλλά δεν μπορούσε σήμερα να παρευρεθεί στη συνεδρίασή μας. Η κυρία Χίεντε ε, θα λάβει λοιπόν το λόγο. Είναι η αρμόδια συγγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να θα σας ευχαριστήσω από πλευράς μου και από πλευράς της κυρίας Μπάουερ για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και σήμερα έχουμε ένα έγγραφο που είναι καλύτερο ουσιαστικά από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατοχυρώνεται με καλύτερη προστασία των θυμάτων, αυξημένες κυρώσεις για τους δράστες. Είναι πάρα πολύ καλύτερο το κείμενο πλέον και είμαστε ευγνώμονες ε, για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε με τους σκιώδεις εισηγητές ε, και με το προσωπικό των επιτροπών. Θα ήθελα να περάσω στα αγγλικά τώρα για να αναφερθώ σε κάποια βασικά ζητήματα. Τα λέω στα αγγλικά γιατί δεν είμαι σίγουρη αν θα με καταλάβετε. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσετε ότι το κείμενο ε, μαζί με τις ε, προσθήκες είναι ένα πακέτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν το το κείμενο του άρθρου 54 τροποποιηθεί όπως προτείνουν οι, προτείνουν οι φιλελεύθεροι με ξεχωριστή ψηφοφορία, τότε θα καταπέσει το σύνολο του πακέτου. Και αυτό θα είναι κρίμα γιατί εργαστήκαμε πολύ σκληρά για αυτό το πακέτο ξεχνάτε, ακόμα και αν περάσουν οι τροπολογίες των φιλευθέρων, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Στο συμφωνημένο κείμενο δεν προβλέπεται καμία δέσμευση ε, των κρατών μελών να ποινικοποιήσουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε αυτό να το ψηφίσουμε αν μπλοκ και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ζητήσατε το λόγο. Θέλετε να κάνετε κάποια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ παρεμβαίνω συντηνιστή της, ε, του ΕΛΚ για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Όπω είπατε η κυρία Μπάουρ δεν είναι εδώ, είναι στο Κονγκό σε μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπή και δεν μπόρεσε να έρθει εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα τη εμπορία των ανθρώπων. Και ε, θα ήθελα να συγχαρώ και τη δική μα τη συνάδελφο, την κυρία Μπάουρ, η οποία κατέβαλε μεγάλε προσπάθειε για αυτό το θέμα και είναι κρίμα που ε, δεν μπόρεσε να είναι κοντά μα σήμερα. Συμφωνώ επίση με την κυρία Χέτ για αυτά τα οποία είπε σχετικά με αυτό το κείμενο ε, και το οποίο εκπροσωπεί εξάλλου και τη θέση ε, του ΕΛΚ. Ευχαριστώ λοιπόν και τους δύο συγητές για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να ακούσουμε και το Συμβούλιο τώρα. Κυρία Γιάνσεν, έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την Βελική Προεδρία, διότι πρόκειται για μία από τι προτεραιότητε του προγράμματό μα και συνιστά προτεραιότητα και για το Συμβούλιο. Έγιναν εντατικότατε διαπραγματεύσει με τι δύο συνεισηγήτρε. ευχαριστούμε παρεμπιπτόντω για τη συνεργασία. Ε, η ένταση των διαπραγματεύσεων με τις συνεισηγήτρες ήταν στο ύψος ε, της σημασίας που έχει αυτή η οδηγία. Μετά τον τριμερή διάλογο, τον τελευταίο τριμερή διάλογο, η Κορεπέρα έδωσε τη συγκατάθεσή της για το κείμενο που σας υποβάλλουν οι συνεισηγήτριες σήμερα και θεωρούμε ότι είναι πλέον ισόρροπο το κείμενο και θα επιτρέψει μετά την εφαρμογή να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον κύριο Μπορατίνσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Εξ ονόματος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας ικανοποίηση για το ότι το Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, την πρώτη οδηγία για το ουσιαστικό ποινωτικό δίκαιο όπου συμμετείχε το Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και δράτουμε την ευκαιρία για να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για αυτή τη θαυμάσια ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε και την πολύ καλή δουλειά των εισηγητών. Για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μια καλή αρχή για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για την ψηφοφορία και για αυτή την πρόταση οδηγίας. Κατόπιν αιτήματο θα κάνουμε ε, ξεχωριστή ψηφοφορία για το 15-4. Τροπολογία 228, 228. Με ανάταση χειρός ψηφίσμου, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για το τελικό κείμενο στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται και η τελική ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. The same Mrs. Yes. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 51 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος κατά συγχαρητήρια. Το Δεκέμβρη θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια και πριν ε, κηρύξω τη λήξη της ε, κοινή συνεδρίασης των δύο επιτροπών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολόθερμα και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αγαστή συνεργασία που έγινε ανάμεσα στις δύο επιτροπές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αγγουλάρ, τον πρόεδρο της Επιτροπής, και τις δύο συνεισηγήτριες ε, θα διαβιβάσω τα καλά νέα και στην κυρία Μπάουερ που αποσιάζει ένα θερμό ευχαριστώ επίσης προς τις δύο γραμματείες των επιτροπών που συνέβαλαν ουσιαστικότατα στην αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων και ευχαριστώ τέλος ε, τα μέλη και των δύο επιτροπών γιατί έδειξαν ιδιαίτερη αφοσίωση και ήταν καταπληκτική η έκβαση της ψηφοφορίας ως εκ τούτου ένα θερμό ευχαριστώ προς όλους όσους συνέβαλαν στις εργασίες. Εμείς θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας στην Επιτροπή Γυναικών.